πρακτικά Έχω δύο ανακοινώσει ακόμα να σας κάνω. Ο κύριος Βλάντιμι Ρέμεκ με ενημέρωσε ότι παρετείται από τις 16 Δεκεμβρίου από τη θέση του Ευρωβουλευτού σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού διαπιστώνει τη χειρία το Κοινοβούλιο από τις 16 12 και θα ενημερώσει σχετικά για αρμοδίως τις ε, αρχές. Ο κύριος Νταν Γιώργερσεν στις 12-12 του διορίστηκε ε, Υπουργός ε, ε, Γεωργίας, Διατροφής και Αλληλίας. Τον συγχαίρω για την ανάλυση των καθηκόντων του. Στις του λοιπόν διαπιστώρεται η χειρία της έδρας του και θα ενημερωθούν οι αρμόδιες δανεικές αρχές. Συζητήσει επί περιπτώσεων παραβίαση τώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου, διάρκεια μία ώρα κατανότητα το όριο,